συζήτηση για τα θέματα αυτά. Τώρα, για τους ανθρώπινους πόρους, νομίζω ότι αυτό είναι άκρα σημασία. Θα πρέπει η επιστήμη, η έρευνα να ενισχύονται διαρκώς και αυτό με μια, ένα σύνολο προσπαθειών από κάθε χώρα. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Και ο κύριο Έλερ και η κυρία Μαντουρέλ τα έφτιαξαν τα ζητήματα αυτά. Είναι προβληματισμοί που και εμά μα φαίνονται πολύ σημαντικοί. Ο κεντρικό χαρακτήρα, τώρα, η κεντρική δομή. Θεμελιώδου σημασία και αυτό. Θα πρέπει να πετύχουμε να έχουμε ένα μέσο, ευρωπαϊκό μέσο, το οποίο να καλύπτει τις ανάγκες της Ευρώπη όλων, τι κοινέ ανάγκε τη Ευρώπη. Και για τα νέα κράτη-μέλη και για τι χώρε του Νότου, θα πρέπει να μην υπάρξει είτε διακριτική μεταχείριση είτε παραγωνισμός σε σχέση με τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης για την έρευνα και την καινοτομία ως προς την απλούστευση. Και αυτό το ζήτημα νομίζω εδώ έχουμε μια κοινή προσέγγιση γενικευμένη και τέλος για τα προβλήματα που εντόπισε η συνάδελφος Ριέρα Μαντουρέλ. Και εγώ θέλω να μοιραστώ μαζί σας το, γεγονό γεγονός ότι είναι σημαντικό τι θα γίνει με τις κοινωνικές επιστήμες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Την ενίσχυση της βαρύτητας που έχουν και το τι γίνεται με τις υποτροφίες των διαφορών ε, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Το πρόγραμμα Μαρή Curie, το οποίο ανέφερε και η συνάδελφος Καρβάλιου, είναι κάτι που θα πρέπει να μας δώσει ένα παράδειγμα για τον ελάχιστο κοινό παρανομαστή των ε, χρηματοδοτήσεων. Όχι περικοπέ, λοιπόν, αύξηση για το... Ευρωπαϊκό λοιπόν Ινστιτούτο Καινοτομία και Τεχνολογίας. Εδώ είναι πολλά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την τροποποίηση του κανονισμού, όπω είπε ο συνάδελφο Λάμπερτ, και αμέσω θα πρέπει να στραφούμε στη διάρθρωση. Την πολύ ξεκάθαρη διάρθρωση για, τον κατάλογο προτεραιοτήτων της καινοτομία με την ε, αυτή καθευτή λειτουργία του Ινστιτούτου. Θα πρέπει δηλαδή από την αρχή να σχεδιάσουμε πώς θέλουμε να διαρθρωθούν οι αρμοδιότητες ε, του Ινστιτούτου, το Ινστιτούτο, οι στόχοι που θα επιλεγούν για το Ινστιτούτο, οι φορείς που θα συμμετέχουν και στις επενδύσεις και στη λειτουργία του Ινστιτούτου με τρόπο ισόρροπο. Όλα αυτά πρέπει να έχουν σχεδιαστεί. Πώς μάλιστα θα λειτουργεί με στόχο την εκπλήρωση των ε, δεσμεύσεων της ε, ατζέντα για την καινοτομία. Βέβαια, πέραν αυτών, θα πρέπει να θέσουμε μία σειρά ερωτημάτων δεν μπορεί να βλέπουμε πάντοτε κοντόφθαλμα το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομία και Τεχνολογία. Θα πρέπει να δούμε το θέμα πιο γενικευμένα, με έναν τρόπο πιο ευρύ, λιγότερο περιορισμένο. Και τι εννοώ με αυτό. Θέλουμε κάτι ισοδύναμο με αυτό που ανέφερε η συνάδελφος Καρβάλιου με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα ή να έχει καταλητικό ρόλο το Ινστιτούτο αυτό ώστε να εξυγχρονιστούν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ανά την Ευρώπη. Δεν θέλουμε να είναι ακριβώ ένα καταλήτη για τον όλο εξυγχρονισμό που επιχειρείται. Για την αριστεία σε όλου του τομεί και στην έρευνα και στην ε, καινοτομία. Θα θέλαμε, θα θέλαμε να το χρησιμοποιήσουμε λοιπόν το Ινστιτούτο κατά αυτόν τον τρόπο ή όχι. Αυτό πρέπει να σκεφτούμε. Και έπειτα για την ευελιξία το πώς μπορεί να γίνει πιο ευέλικτος ο τρόπος λειτουργίας του. Εδώ λοιπόν πρέπει να πρικοδοτήσουμε με ένα τέτοιο βαθμό ευελιξία το Ινστιτούτο στον τρόπο λειτουργίας του και πώς θα συσχετιστεί αυτό με άλλες παραμέτρους της λειτουργίας, της χρηματοδότησης, λιγότερη απόδοση αρμοδιοτήτων, ε, λιγότερη λογοδοσία, είναι αυτό που, επιτέχ που επιθυμούμε. Έχουμε αρκετέ γνώσει, νομίζω, αρκετή πείρα από τη λειτουργία του Ινστιτούτου, αρκετά πρόσφατα πορίσματα και αρκετά πρόσφατο έργο για να μπορέσουμε να βασιστούμε και να δούμε τι θέλουμε μεταξύ των δυνατοτήτων ανάπτυξης του Ινστιτούτου και του καλύτερου σχεδιασμού του, με μεγαλύτερη σαφήνεια μάλιστα. Εκεί θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας. Και έπειτα υπάρχει και μια πολύ συγκεκριμένη διάσταση που έχει σχέση με αυτό που πραγματικά κάνει τη διαφορά. Είδαμε πώ συμμετέχουν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ω τώρα, τα ερευνητικά ιδρύματα, ο ιδιωτικό τομέα τη βιομηχανία. Υπάρχει ένα τρίγωνο λοιπόν συνεργασίας, το οποίο διαρκώς εξελίσσεται. Οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειακοί, τοπικοί φορείς, πολύ σημαντική και αυτή η διάσταση. Μπορούμε να την επεξεργαστούμε περαιτέρω, να εμβαθύνουμε στην διάσταση των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης. Όμως τι είναι αυτό που διαφοροποιεί πραγματικά το Ινστιτούτο. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με την εκπαίδευση, με την κατάρτιση. Δηλαδή αυτό που είναι το κοινό στοιχείο όλων των εκθέσεων, όλου τις δέσμες προτάσεων, μιλάνε φυσικά για την έρευνα, για τις κατευθύνσεις της αριστείας, για τις προκλήσεις, τις κοινωνιακές, τις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις, αλλά εμείς θέλουμε να δούμε τι συμπληρωματικά στοιχεία υπάρχουν, αλλά και τι διαφοροποιεί τα διάφορα στοιχεία του ορίζοντα 2020 δεν μπορεί να είναι ούτε γιγαντιαίων διαστάσεων, τιτάνιων αυτό το πρόγραμμα, αλλά ούτε και μικρό, νάνος. Θα πρέπει λοιπόν εδώ στην καινοτομία να επεξεργαστούμε με πολύ προσοχή το στοιχείο αυτό και ιδίως το Ινστιτούτο. Έχοντας ακούσει τώρα τις απόψεις των συναδέλφων, πιστεύω ότι θα χρειαστούν ακόμη πολλές, πολλές, πολύ συζητήσεων για να αποσαφηνίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα, όλες αυτές τις προτάσεις. Πάντως, η καινοτομία μπορεί να προαχθεί από το Ινστιτούτο. Για τον κεντρικό χαρακτήρα τώρα που θέλουμε να δώσουμε στη διάρθρωση του συστήματος, μια ανησυχία που μπορεί να έχουμε εδώ είναι ότι νέες τάσεις θέλουμε να έχουμε, νέες ιδέες. αλλά θα θέλαμε το Ινστιτούτο να είναι και ένα στοιχείο που να ενώνει τις διάφορες περιοχές της Ευρώπης, ακόμα και τις μακρινές ακόμα και, και τις κεντρικές. Θα μπορούσε να γίνει ένας παράγοντας ε, που να προάγει την Ευρωπαϊκή Συνοχή από αυτή την άποψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την συνάδελφο Ματίας και τώρα ακούμε τις παρεμβάσεις των υπολείπων συναδέλφων. Έχω 11 αγορητές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε με τη συνάδελφο Γκουτιέρες Κορτίνες για δύο μισή λεπτά. Ευχαριστώ. Α, ο κύριος Έλερ προηγουμένως. Ε, θα είχα μια ερώτηση. Ορίστε, αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα της συζήτησης. Εγώ ως εισηγητής θα ενδιαφερόμουν πάρα πολύ να ακούσω τη θέση των ε, σκιωδών εισηγητών, συγκεκριμένα των σοσιαλιστών και δημοκρατών για τη δική μου έκθεση. Βεβαίως ε, συζητήσαμε κάποια πράγματα μεταξύ μα, αλλά επειδή θέλουμε να έχουμε συλλογική προσέγγιση, καλό θα ήταν να ε, ακούμε τον εισηγητή και τους σκιώδη για όλες τις εκθέσεις. Καλό είναι να έχουμε κατάλογο μιλητών, αλλά ε, δεν υπάρχει σωστή διάρθρωση, δεν λειτουργεί καλά αν δεν ανταλλάσσουν απόψει οι σκιώδη με τους εισηγητέ. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Ελέρ που μου δίνει την ευκαιρία να κάνω μια επεξήγηση. Είναι τρει και ο στη σειρά που έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κύριο Φόρντ, ο κύριο Φανίστε Ρόι και ο κύριο Τζόνσον. Μέχρι τώρα αυτοί οι συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο από του ο εισηγητέ. Οι υπόλοιποι δεν έχουν γραφεί. Εάν Μπορεί να παρέμβει όμω ο συνάδελφο που σα είπα προηγουμένω, γιατί είχε ζητήσει το λόγο πριν ακόμα από την αρχή τη συνεδρίαση. Θα έλεγα λοιπόν να είχαμε την ευγενή καλοσύνη να τη επιτρέψουμε να κάνει την παρέμβασή του τώρα για δύο λεπτά. Για την κυρία Γκουτιέρε δηλαδή. Και μετά θα περάσουμε στου σκιώδει εισηγητέ. Τρει έχουν αγραφεί όπω σα είπα, μόνον. Αλλά θα του ακούσουμε έτσι κι αλλιώ. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ Πρέπει να ε, πάω να συναντήσω έναν επίτροπο και δεν προλαβαίνω, γι' αυτό πρέπει να φύγω. Πολύ σύντομα. Εδώ και πολύ καιρό εγώ μελετώ το πρόγραμμα αυτό και μάλιστα το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και έψαξα να δω τι έγινε στο 7ο. Και εγώ ανησυχώ πάρα πολύ περισσότερο εάν το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνεχίζει τα προβλήματα ή τις ελλείψεις του 7ου προγράμματος πλαισίου δεν θέλω να πω ότι είναι μελανά τα σημεία γιατί είναι αρνητικό όρο, αλλά είναι πολλά τα κενά από το προηγούμενο πρόγραμμα πλαίσιο. Προσπαθεί το πρόγραμμα να δώσει κάποια συνοχή, να συμπεριλάβει κάποια θετικά θέματα. Δεν θέλω όμως η παρέμβασή μου να είναι αμυγός επενετική. Να σας πω τα προβλήματα που έχω εντοπίσει. Συμφωνώ απολύτως με την κυρία Ριέρα. Το πρόβλημα των ανθρωπίνων πόρων παραμένει ανεπίλητο και μάλιστα έχει επιδεινωθεί. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε αποκέντρωση, η οποία δεν ήταν γεγραμμένη, αλλά έγινε από τον κύριο Μπαρόσο, χωρίς να συνεννοηθεί με κανένα, το αποφάσισε ο κύριο Μπαρόσο και πολλά από τα προγράμματα αποκεντρώθηκαν σε άλλες γενικές διευθύνσεις που δεν είναι Γενική Διεύθυνση Έρευνα. Έχουμε μεγαλύτερο καταγερματισμό. Λοιπόν, επιπλέον, απαγκίστρωσε το Marie Curie από το πρόγραμμα της έρευνας. Και αυτή η ιδέα που επικρατούσε από την αρχή ότι ε, πολλές υποτροφίες πηγαίνουν σε συγκεκριμένα προγράμματα έχει διαταραχθεί αυτό. Εάν θέλουμε οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν, πολλοί υπότροφοι θα πρέπει να εκπαιδεύονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αυτό κάνει η Γερμανία, για παράδειγμα, και με διδακτορικά και στην Αμερική. Δεν το λαμβάνουμε υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ανθρώπινη πόρη, συγγνώμη, δεν είναι επαρκής. Δεν έχουμε ερευνητές στην Ευρώπη. Οι Ηνωμένε Πολιτείε στρατολογούν από την Ασία και από άλλες περιοχές, εμείς όχι. Επίσης με ανησυχεί πολύ γιατί αυτή η αποκέντρωση δημιούργησε μια δυσκολία στον έλεγχο και τον ποιοτικό έλεγχο και τη συνοχή. Υποπτεύομαι ότι στη Γενική Διεύθυνση Έρευνα θα πρέπει να επικρατεί μεγάλη απογοήτευση για το λόγο αυτό. Στο πρώτο παράδειγμα, το κεφάλαιο για την αριστεία είναι πολύ περιορισμένο. Νομίζω πρέπει ο όρος αυτός να τύχει περισσότερης επεξεργασίας και επεξήγησης. Έχουμε τεράστιες δυνατότητες στο πρόγραμμα, αλλά χρειάζεται συντονισμός. δεν έχουμε διερευνήσει ε, ε, τα κοινά προγράμματα, το joint ε, program. Θα τα δούμε βέβαια αυτά στα ειδικά προγράμματα, αλλά ακόμα υπάρχει χώρος εκεί για περισσότερη διερεύνηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Κουτιέρες. Φόρτ, παρακαλώ. Hi, it's Mrs. Ford. Um, thank you. I'll try and be quick. Um, Ευχαριστώ. Είναι κυρία Φόρτ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Άκουσα τα σχόλια τη κυρία Γέρα Μαντουρέλ, τα οποία βρήκα πολύ διαφωτιστικά, για το μέγεθο του προπολογισμού συμφωνώ με τον κύριο Έλερ. Πρέπει να το συζητήσουμε μαζί με το MFF. Πρέπει να δούμε το συνολικό πλαίσιο τη χρηματοδότηση δηλαδή. Τώρα για τον ισόρροπο προπολογισμό. Μιλήσατε για τη μακροπρόθεσμη έρευνα και το πώ αυτό θα πρέπει να εξισορροπηθεί σε σχέση με την πρόθεσμη έρευνα. Αυτό απομένει να το συζητήσουμε για τους ε, βασικούς στόχους, τους ε, κεφαλαιώδεις στόχους. Καλά είπε ο κύριος Λάμπερτς ότι αυτούς θα πρέπει να τους ε, μελετήσουμε από κοινού, αλλά λόγω χάρη αν έχουμε κάποιο στόχο για διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας μερικές φορές καθυστερούν και οι ιδέε, ε, οι ανακαλύψει μεταδίδονται διαφορετικά μεταξύ των επιστημόνων. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το σκεφτούμε για το θέμα τη αριστεία. Συμφωνώ με όσα υπόθηκαν, ιδίω από την κυρία Καρβάλιου. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η αριστεία θα απλωθεί και στου τρει πυλώνε και επίσης να δούμε την συμμετοχή, λόγου χάρη τη βιομηχανική ηγεσία. Ναι, σε αυτόν τον πυλώνα θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, λόγου χάρη. Και όντω πρέπει περισσότερο να εμβαθύνουμε για την για το πώ συσχετίζονται με τα δημοσιοτικά ταμεία οι προσπάθειε αυτέ περί αριστεία για το θέμα τη συμμετοχή. Όντω, πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να κινητοποιηθεί και ο ιδιωτικό τομέα. Άρα, μέρο τη συμμετοχή, ιδίω για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, είναι καιρό να δούμε ότι θα πρέπει κάποιε φορέ να πληρώνεται ε, θα ήθελα να μιλώ εγώ εφόσον είναι η σειρά μου. Ε, την, την προηγούμενη φορά στην Ευρωπαϊκή, ρωτήσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τρει επιτρόπου τι γίνεται με την συμμετοχή των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ένα πρόγραμμα που ακόμη περιμένει το κονδύλι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι τρει επιτροποί πριν δέκα μέρε έλαβαν τα, ε, το ερώτημά μα και δεν έχουμε λάβει εμεί καμία απάντηση. Μεγάλε καθυστερήσει λοιπόν με τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για το Ινστιτούτο, συμφωνώ με την αύξηση του χρηματοδότου τη χρηματοδότησή, όμω δεν ξέρω κατά πόσο θα υπάρξει δυνατότητα απορρόφηση με το πρόγραμμα IT. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε ότι αν το Ινστιτούτο μπορεί να απορροφήσει τα κονδύλια με τρόπο που να αποδίδουν και ω προ το κόστο. Και επίση διαφορετικέ πηγέ επιστήμονε ή ε, επιστήμες. Ε, ε, εδώ μας έκανε εξαιρετική πρόταση η κυρία καρβαλιο το κόστο του εξοπλισμού λόγω χάρη θα μπορούσε να καλύπτεται από το άμεσο κόστο αυτό. Θα μπορούσε να επιλύει ένα μέρο του προβλήματο. Εάν όχι, να δούμε τι γίνεται με το πραγματικό κόστο για τη μεγαλύτερα ερευνητικά ιδρύματα ή τι οργανώσει. Αυτό νομίζω θα μπορέσουμε να το επεξεργαστούμε με τον κύριο Έλερ, να δούμε τι λεπτομέρειε των κανόνων συμμετοχή εδώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Τζόνσον. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ είμαι σκιώδη συγητή ε, από πλευράς φιλελευθέρων και έχω κάποιες παρατηρήσεις που μπορεί να σα φανούν χρήσιμες σε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Καταρχάς, θα πρέπει να γίνει μια ανοιχτή συζήτηση ε, μεταξύ των ε, εισηγητών και των σκιωδών εισηγητών. Τη θεωρώ χρήσιμη και σκόπιμη. Βλέπω ότι γενικά στην Επιτροπή μας υπάρχει συναντήληψη για αυτά τα θέματα. Να σας πω τι λέει η πολιτική μου ομάδα. Πρώτα απ' όλα για τα δημοσιονομικά. Θεωρούμε και εμείς ότι θα πρέπει να προσανατολίζεται ο προϋπολογισμός προς την έρευνα και την καινοτομία φυσικά Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχαμε με τους συναδέλφους της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμών και της ε, Περιφερειακής ε, Πολιτικής διαφάνει σε ποιο βαθμό μπορούν αυτά τα προγράμματα να συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων για το 2020. γιατί ακριβώς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις τις οποίες ζούμε. Ένα άλλο σημείο που θέλω να αναφέρω εκτός από τον προπολογισμό είναι να υπάρχουν περισσότεροι συμμετέχοντες και αυτό συνδέεται και με τα διορθωτικά ταμεία και την πολιτική συνοχής. Πραγματικά θα πρέπει να δημιουργηθούν και συνεργασίες και συνέργειες στο παρελθόν είχα ασχοληθεί με τα διαθροτικά ταμεία και τα προγράμματα καινοτομία και μπορώ να σας πω από την πείρα μου ότι υπάρχουν δυνατότητες ακόμα συνεργασίας και μπορούν να συμβάλλουν τα διαρθρωτικά ταμεία. Ακριβώς να δημιουργήσουμε τέτοιες δομές συνεργασίας που να προωθούν και την καινοτομία και την έρευνα και την αριστεία στην έρευνα. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό. Και τα νέα κράτη-μέλη να συμμετέχουν με τρόπο πιο εντατικό στην έρευνα και στην ε, καινοτομία. Και όχι μόνο τα νέα μέλη αλλά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και περισσότερο οι γυναίκες ερευνήτριες ε, στην έρευνα και την καινοτομία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας είναι καλό να δραστηριοποιηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Αλλά συμφωνώ και με τις ερωτήσεις των συναδέλφων και με τις αμφιβολίες τους. Υπάρχει δυνατότητα καν απορρόφησης, υπάρχουν αυτές οι δομές. Το πρόγραμμα χρειάζεται απλούστευση και μείωση της γραφειοκρατίας για να μπορέσουμε πραγματικά να φροντίσουμε να συμμετέχουν καλύτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μπορεί να υπάρχει παγκοσμιοποίηση και μεγάλες εταιρείες. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η έρευνα και η καινοτομία να μπορεί να γίνεται και στις μικρές και μισές επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Έλερ. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω το χρόνο μου πολύ γρήγορα διότι έχουμε σαν προσκεκλημένο τον Γενικό Διευθυντή και δεν θέλω να του φάω το χρόνο του. Αλλά καταρχήν σχετικά με τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Νομίζω ότι ίσως ε, υπάρχει ε, ένα συγκεκριμένος ορισμός στον χώρο αλλά δεύτερον ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορα Ινστιτούτα, Think Tank, το CRC τι, πώς βλέπετε να εξελίσσετε το GRC στο μέλλον και ποια θα είναι τα βασικά του καθήκοντα. Το τρίτο αναφέρεται στην καινοτομία, το οποίο ανέφερα προηγουμένως. Δηλαδή, μέχρι στιγμής το πρόγραμμα είναι σε πυλώνες και ε, είναι ε, σαν ε, τη συνήθη ροή. Ζητούμε ένα πρόγραμμα στο οποίο θα συμμετάσχουμε και υπάρχει, συμβαδίζει και με την καινοτομία. Αλλά υπάρχει και ένα ενδιάμεσο στοιχείο μεταξύ της έρευνας και της επιστήμης, δηλαδή ένα καινοτόμο πρόγραμμα και η Επιτροπή μας είπε ότι θα υπάρχει ένα ευρύ πεδίο μεταξύ της έρευνας και της καινοτομίας αλλά το θέμα είναι πώς θα ζητούμε αυτό που θέλουμε δηλαδή πώς το πρόγραμμα θα απομονώνεται η καινοτομία θα είναι ένας πυλώνας ο οποίος ε, θα μας, ε, στον οποίο θα ζητούμε συγκεκριμένα θέματα ή η καινοτομία δεν θα είναι ένας ένας αλλά ένα οριζόντιο θέμα σε ένα πρόγραμμα όπου το θέμα της καινοτομίας θα είναι ένα θέμα του συνολικού προγράμματος. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί. Ε, πέραν ε, της θεωρίας και της σκέψεως πρέπει και στην πρακτική να το χρησιμοποιήσουμε για να πετύχουμε και όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία. Είναι κάτι που έχουμε συζητήσει πολύ και θα αναλάβουμε και προτάσεις, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, το έχει επεξεργαστεί. Δηλαδή, μεταξύ αυτών τα οποία λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα διαρθρωτικά ταμεία και για το πρόγραμμα Horizon, πόσο θα υπάρξει μία διασύνδεση και πού θα παραμείνουν οι αρμοδιότητες ε, του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ κύριος Βανίστερόι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σύντομα κάποιες σημειώσεις. Τα θετικά τα είπε η κυρία Μαντουρέλ και τα γράφει και στην έκθεσή της. Είναι οι τρεις πυλώνες και πώς συνεχίζεται αυτή η διάρθρωση σε δύσκολους καιρούς, ε, χαλεπούς καιρούς και κρίση. Κάθε ευρώ θα πρέπει να πιάνει τόπο. Ε, λοιπόν, ποια είναι η θέση της καινοτομίας και αν έχουμε την αριστεία ως αφετηρία θα πρέπει να το διατηρήσουμε. Το βλέπουμε αυτό στη θεμελιώδη έρευνα, στην εφαρμοσμένη έρευνα και εκεί σταματάει. Αν αυτό δεν μπορείτε να το μεταβιβάσετε στην πραγματική ζωή, στις εταιρείες, στη χώρα σας, στις περιφέρειες, παντού στην Ευρώπη, είναι σφάλμα. Ε, θα πρέπει να επιλέξετε στο πρόγραμμα ορίζων ε, πώς θα τονωθεί η ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη και η κατάρτιση και η εκπαίδευση ε, των Ευρωπαίων. Η τέχνη αυτή είναι πραγματικά να μπει στην αλυσίδα του ορίζοντα ε, και ο κόσμος και να συμμετέχει η πραγματικότητα. Να πω για την αριστεία λοιπόν ακόμα κάτι διαβάζοντας τα έγγραφα διαπιστώνει κανείς ότι είναι πάρα πολύ ασαφή και συγκεχημένα και αόριστα. Το είπε και ο κύριος Έλερ. Και θα πρέπει να σκεφτούμε τι κάνει κάθε χώρα στην εταιρική σύμβαση από το 2013 και μετά. Ε, Δεσμεύσει δηλαδή μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών που ε, κάνουν χρήση των διαφορετικών ταμείων και δεσμεύονται τι θα κάνουν. Εκεί βλέπετε ποια κράτη-μέλη, σε ποια πόλη, σε ποια περιφέρεια, με ποια πανεπιστήμια ποντάρει στην ευφυή e e εξειδίκευση, smart specialization. Και από εκεί και πέρα ε, αφήνουμε τους γενικούς κανόνες και μπορεί η χώρα Α να επιλέγει μια κλασική υποδομή. Ας είναι. Μια άλλη χώρα Β επιλέγει πιο πολύ για έρευνα και υποδομές. Εκεί χρειάζεται μια κοινή διαχείριση, share management, μεταξύ ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων. Εκεί υπάρχουν πολλές ε, δυνατότητες. Το ε, ε, EIT χρειάζεται μετεξέλιξη, όχι επανάσταση. Η Επιτροπή μας, η ΤΡΕ, δεν είχε πει ποτέ ότι χρειάζεται επανάσταση. Εμείς θυμάστε γίναμε περίελος, μας κλέβασαν όταν είπαμε ότι θέλουν να συμμετέχει και βιομηχανία. Μπορεί τα πρώτα χρόνια να υπάρχουν δυσκολίες, αλλά πραγματικά και στα ΚΙΚΣ και στις άλλες πρωτοβουλίες ε, θα πρέπει να βλέπουμε μια αντανάκλαση της πραγματικής οικονομίας και της πραγματικής βιομηχανίας. 50% χρηματοδότηση μπορεί να είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 50% από την ιδιωτική βιομηχανία. Γιατί όχι θα πρέπει να προσελκύσουμε επενδύσεις. Το να μοιράζουμε δεξιά και αριστερά λεφτά, αυτό τα κάνει μόνο ο Άγιος Βασίλης. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε εμείς και να είναι και το μέλλον μας αυτό και η ιδεολογία μας για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Τσουκαλάς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ χρήσιμη συζήτηση και είναι προφανές ότι όλοι οι συνάδελφοι υποστήριξαν ε, τις απόψεις τους πάνω σε κείμενα που ο κύριος Βανίστερ Λόι μόλις τα χαρακτήρισε αόριστα. Αυτό συμβαίνει για ένα πολύ απλό λόγο. Οι συντάκτες αυτών των εξαιρετικών κειμένων έχουν μπροστά τους τα συγκεκριμένα στοιχεία που βάζουν την Ευρώπη στο παγκόσμιο σκηνικό. Δεν νομίζω για παράδειγμα ότι αποτελεί κοινή γνώση των συναδέλφων ποια είναι η θέση της Ευρώπης στο παγκόσμιο σκηνικό. Ακούν διαδόσεις, ακούν αποσπασματικά στοιχεία. Για παράδειγμα, είμαστε πρώτοι, είμαστε τελευταίοι, η στρατηγική της Λισαβόνας απέτυχε, πέτυχε, τι έκανε. Θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον πριν αρχίσουμε αυτές τις συζητήσεις μια που έχουμε σήμερα το προνόμιο να έχουμε και το Γενικό Διευθυντή της έρευνας, είτε με ένα κείμενο εργασίας που δεν χρειάζεται να έχει όλη τη σοφία του κόσμου. Αλλά όμως θα ήθελα να ξέρω. 1,33 είναι η παγκόσμια ετήσια μπίζνα για την έρευνα και την ανάπτυξη. Ξέρουμε πόσο συμμετέχει η Ευρώπη σε αυτό ξέρουμε ακριβώς ποια είναι τα ισχυρά μας στοιχεία. Ακούω να γίνεται μεγάλη κουβέντα για τα κίξ. Ε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, έχουμε τρία και θα κάνουμε έξι κίξ και οι Αμερικάνοι έχουν 150. Δεν τα λένε knowledge και information communities, τα λένε regional innovation communities είπε μία συνάδελφος πριν και πολύ σωστά το είπε. Και τι ξέρουμε ότι κάνουν αυτά τα κίξ για τη βιομηχανία. Το είπε και ο κύριος Λάμπερτ πριν από λίγο. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Παράδειγμα το κικ, το, το ρικ που είναι στο Κάνσας και ασχολείται με την αεροπορία έχει το 20% της τοπικής απασχόλησης με μέσο μισθό 65.000 δολάρια όταν η μέση αμοιβή της περιοχής είναι 45.000 δολάρια αυτά κάπως συμμαζεμένα θα έπρεπε να τα μάθουμε. Και θα έπρεπε να τα μάθουμε γιατί δεν έχω καμία απολύτως εμπιστοσύνη ούτε στα οράματα όπως λεγόταν πριν από δύο χρόνια ο Horizon 2020 τότε ήταν Vision τώρα είναι Horizon αν δεν μου εξηγήσει κανείς που είμαστε θα μου εξηγήσει κανείς παραδείγματι εάν το impact που έχουμε στην αγορά είναι αυτό που έπρεπε να έχουμε. Άρα θα πρότεινα, θα παρακαλούσα κυρία Πρόεδρε και με τη δική σας παρέμβαση αυτό να γίνει. Thank you, Chair. Ευχαριστούμε, συνάδελφος Μέρκης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους εισηγητές, τη βασική εισηγητρία μάλλον για το εξαιρετικό έγγραφό τη και τους υπόλοιπους συναδέλφους ότι, για την εμπιστοσύνη τους ότι όλη αυτή η προσπάθεια θα είναι επιτυχής. Και εγώ έχω την αυτοπεποίθηση ότι θα επιτύχουμε εδώ. Όμως τα καθοριστικά ζητήματα, το, το βασικό ζήτημα μάλλον, είναι ότι πρέπει να κάνουμε επιλογές. Θέλουμε αριστεία, θέλουμε συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θέλουμε και κοινοτομία, θέλουμε και αγορά να λειτουργεί, Θέλουμε να εξεύρουμε λύσει για τι μεγάλε κοινωνιακές προκλήσει. Όμω αυτό είναι και ο φόβο μα, ότι αν τα θέλουμε όλα, μπορεί τελικά να καταλήξουμε να μην πετύχουμε τίποτα. Πρέπει λοιπόν να γίνουν επιλογέ. Εάν δούμε τον κατάλογο προσδοκιών των μεν και των δεν, όλοι θα σα πούν ότι πρέπει να γίνουν κάποιε επιλογέ. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό, ιδίω σε αυτή τη χρονική φάση. Υπάρχουν λοιπόν ε, τρία ζητήματα. Προτεραιότητε, σχέσει συνεργασία και να ε, καθορίσουν τις προσπάθειές μας τα αποτελέσματα, κατά προτίμηση τα μετρήσιμα αποτελέσματα. Μίλησα πολύ για το θέμα των επιλογών. Να σταθώ και στο εξής. είναι προτεραιότητα το να επιλέξουμε έξι μεγάλες κοινωνιακές προκλήσεις. Σε όλες τις εκθέσεις, αν σωστά θυμάμαι, η Ένωση για την Καινοτομία μας λέει ότι θα πρέπει να επιλέξουμε τρεις προκλήσεις. Και ό,τι και αν κάνουν ε, στα πλαίσια αυτής της Ένωσης ε, ελέγχονται βάσει αυτών των τριών προτεραιοτήτων. Ίσως πρέπει λοιπόν να μειώσουμε τι πολλαπλές προσπάθειε, να αναζητήσουμε εδώ ακριβώ τη σχέση συνεργασία. Ναι, θα πρέπει να είναι οριζόντιο αυτό το ζήτημα, θα πρέπει να βρίσκεται παντού η καινοτομία. Είναι λοιπόν τώρα η στιγμή να καταλάβουμε ότι καλό είναι να έχουμε περιορισμένε φιλοδοξίε, μάλλον μετριασμένε, να απλουστεύσουμε τα πράγματα και να αναζητούμε σχέσει συνεργασία μεταξύ όλων των ταμείων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των περιφερειακών και των διορθωτικών ή των ταμείων τη κοινή αγροτική πολιτική. Όμω, ε, σχέσει συνεργασία χρειάζονται και μεταξύ των εθνικών πολιτικών, των ε, πολιτικών τη περιφερειακή ανάπτυξη. Υπάρχει και ένα βαθμό σύγκληση εδώ. Ε, το καλύτερο είναι να εκμεταλλευτούμε τι σχέσει συνεργασία που μπορεί να δημιουργούνται. Έτσι θα πετύχουμε αποτελέσματα. Και νομίζω υπάρχει και ένας ακόμη κίνδυνος να μην αναπτυχθούν σχέσεις συνεργασίας μεταξύ όλων των μέσων που διαθέτουμε λόγω χάρη τα ΚΙΚ από το Ινστιτούτο και οι σχέσεις ε, δημόσιου δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Εδώ υπάρχει σε έναν πυλώνα το τι γίνεται με την έρευνα και την υποδομή των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων πολλές φορές ε, κοιτάζουμε το νόμισμα από την μια του όψη, αλλά δεν αλλάζει τελικά η εικόνα, εάν τη δούμε συνολικά. Επίσης, τα αποτελέσματά μας θα πρέπει να είναι μετρήσιμα. Θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές οι προσπάθειές μας, αποδοτικές. Εδώ η τεχνολογία, λόγου χάρη, οι υπηρεσίες ε, τεχνολογίας. Εάν επιλέξουμε τεχνολογικά μέσα θα επιλέξουμε και εργαλεία. Με αυτή τη νέα προσέγγιση, εφόσον επιλέξουμε λόγω χάρη τις μεγάλες κοινωνιακές προκλήσεις, θα πρέπει να επιδιώκουμε ένα τελικό αποτέλεσμα. Αλλά όχι χωρίς επιλογή και το εργαλείο αυτό. Είναι μια σημαντική παράμετρος του ορίζοντα 2020. Θα πρέπει πάντα να το έχουμε κατά νου. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γκλάντε δεν θέλει. No, δεν το Ωραία. Ολοκληρώσαμε τον κατάλογο. Ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των ε, σχεδόν συγκητών. Να δώσω το λόγο σε όλους τους υπόλοιπους. Ο κύριος Τιζέλη. Ε, ευχαριστώ. Απλώς να ενώσω τη φωνή μου με αυτή όλων των υπολείπων συναδέλφων που καλωσόρισαν το πρόγραμμα αυτό. την δέσμη προτάσεων για το ορίζοντα 2020. Είναι καιρός και για απλούστευση και για ανανέωση. Προ προς τον προπολογισμό θα συμφωνήσω με ό,τι είπαν οι συνάδελφοι. 80 δις ευρώ είναι ελάχιστο ποσό. Το ελάχιστο ποσό εάν θέλουμε να πιστέψουμε στο μέλλον της έρευνας εάν θέλουμε να πιστέψουμε στην ανάπτυξη. Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τις προτεραιότητέ μα λοιπόν του ερχόμενου μήνε. Είναι το ελάχιστο ποσό που θα μπορέσει να καλύψει τι ανάγκε μα ε, ο προπολογισμό των 80 δι. Και επιμένω σε αυτό. Όπως ήδη ακούστηκε αρκετές φορές ως τώρα, δεν ομιλούμε μόνο για μεμονωμένα κρατημέλη. Είχαμε μια καθοριστική σημασία συζήτηση στις αρχές του Νοέμβρη και πάλι εδώ και να ευχαριστήσω τον κύριο Σμιθ για την τόσο ανοιχτόμυαλη προσέγγιση του. Ακούσαμε πολλά για τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να εντείνει τα όσα ήδη κάνει, να συμπεριλάβει περισσότερους παράγοντες και φορείς στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, την ενδυνάμωση της καινοτομία και των υποδομών μα ένα τα κάτι μελη Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν περισσότερα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς ε, συμπεριλήφθησαν όλε αυτέ οι προθέσεις στο ίδιο το πρόγραμμα. Κάτι άλλο στο οποίο θέλω να σταθώ. Είναι θα ήθελα περισσότερα στοιχεία για την πρόσβαση, την πρόσβαση αυτή αυτή στα κονδύλια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχετε να μου πείτε κάτι συγκεκριμένο περί αυτού και κάτι άλλο αρκετά συγκεκριμένο επίση. Τα περιφερειακά προγράμματα, ξεκινώντας από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο που μεταφέρονται υπό τη σκέπη των προγραμμάτων συνοχής δεν υπάρχει εδώ και αλλαγή στα κριτήρια για την πρόσβαση στα κονδύλια και τη χρηματοδότηση. Θα ήθελα και εδώ διευκρινήσει. Επίση, κάτι ακόμη. Οι πυλώνε του ορίζοντα 2020. Για τον πυλώνα της έρευνας υπάρχει το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Συμβούλιο. Ακούστηκαν οι μελλοντικέ ε, τεχνολογίες, θα ήθελα, περισσότερο για περισσότερα λόγια για το πώς θα διαχωρίζονται οι ρόλοι αυτών των οργάνων. Διότι θα υπάρξει μια κατανομή του προπολογισμού, αλλά και δωρεές προς κάποια, κάποιους ομίλους. Έχω αυτές τις ερωτήσεις προς το παρόν, αλλά και πολλές ακόμη για επόμενες φάσεις της συζήτηση. Ευχαριστούμε. Κυρία Τερκαστήγιο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια και συγχαρητήρια και στους υπολείπους που έχουν ε, την ευθύνη των εκθέσεων αυτών. Είναι μεγάλο το εγχείρημα για την ανάπτυξη, την έρευνα και την καινοτομία που θα αντικαταστήσει και το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και τα συνοδευτικά προγράμματα. Και πάλι γενική συζήτηση κάναμε τώρα όμως. Κάποια Άλλη στιγμή θα πρέπει να μπούμε σε πιο συγκεκριμένε συζητήσει για κάθε έκθεση ξεχωριστά. Γιατί δεν μπορούμε συνεχώ να συζητούμε επί παντό επιστητού. Επιτρέψτε μου να κάνω κάποιε μικρέ σκέψει, χωρί να επεκταθώ πολύ ε, για τη δομή, για τα μέσα συμμετοχής και για τους κανόνες συμμετοχής. Σε ό,τι αφορά τη δομή και τη διάρθρωση, ακούστηκε και προηγουμένως. αυτό το τρίγωνο της γνώσης, έρευνα, ε, καινοτομία και τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι πολύ ε, εύστοχο και πραγματικά αξίζει ε, συγχαρητήρια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, το Κοινοβούλιο έχει κατά την απόψή μου ακόμα περιθώριο για να διευκρινίσει κάποιες έννοιες σημαντικές. Ας πούμε, το όραμα της στήριξης στην καινοτομία, στο πρόγραμμα και στην πρόταση ορίζον 2020 ε, είναι περιοριστική και ασαφής γιατί δεν κάνει μία διάκριση με την ερευνητική δραστηριότητα γιατί που χρειάζεται να γίνει η συμμετοχή των φορέων ε, στην έρευνα επηρεάζει το ποσοστό επιδότησης που μπορεί να πάρει κάθε χωρέα από το 100% είναι έρευνα και ανάπτυξη, 70% είναι καινοτομία, πρωτότυπα, ε, επιδείξεις κτλ. Από την άλλη, η τριτοβάθμια εκπαίδευση συνδέεται στο τρίγωνο και το γνωρίζουμε κυρίως με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Ιδρύματος. Δηλαδή υποστηρίζουμε ε, τις επιχειρήσεις. Αυτό όμως θα πρέπει να συνοδεύεται από ρητή υποστήριξη των πανεπιστημίων που δίνουν διδακτορικά και ε, τις δράσεις υποτροφής Marie Curie. Σε ό,τι αφορά ε, τα μέσα συμμετοχής, προσοχή. Γιατί υπάρχει μια τάση να δίνεται κάποια προτεραιότητα σε δράσεις και ε, πολύ μεγάλη εμβέλεια και βεληνικού. Εγώ θα προτιμούσα να ενισχύονται μικρά προγράμματα που βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα πανεπιστήμια. Σε ό,τι αφορά τους κανόνες τέλο συμμετοχή, έχουν γίνει μεγάλα βήματα ε, προόδου για την απλούστευση, αλλά ακόμα εκρεμεί μεταξύ άλλων η αύξηση και εγώ θα έλεγα δραστική αύξηση των πληρωμών ε, για έργο που παρέχουν κάποιοι όμιλοι αυτό το μέτρο το αναμένει η επιστημονική και ερευνητική κοινότητα και πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να βοηθήσει και εδώ όπως και αλλού. Έχει αρκετό ε, περιθώριο και μεγάλο ρόλο ακόμα να διαδραματίσει. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κέλλη παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ. Θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ πρακτική, διότι έχουμε τον ορίζοντα 2020, αλλά απέχει πολύ από τα 100 δισεκατομμύρια τα οποία επιθυμούσαμε αρχικά και το πρώτο θέμα που θέλω να θίξω είναι ότι αν θέλουμε να φτάσουμε στο 3% του ΑΕΠ για ε, προπολογισμό, χρειαζόμαστε να εμπλέξουμε ακόμη τουλάχιστον ένα εκατομμύριο άτομα ακόμη. Είμαστε εστιασμένοι για να εξασφαλίσουμε ότι θα εμπλακούν όλοι αυτοί οι πολίτες και επίσης σχετικά με αυτό που είπε ο κύριος Βαλνίστερ Ρόι, πρέπει να υπάρχει διασύνδεξη ε, μεταξύ της έρευνας και της βιομηχανίας. Αλλά η βιομηχανία θα ασχοληθεί με την έρευνα μόνο αν αποκομίσει κάτι. Οπότε τα εκπαιδευτικά ε, Ινστιτούτα, ναι μεν μπορεί να ε, είναι εμπειρογνώμονες ε, σε θέματα ερεύνης που δεν έχουν όμως πρακτικές εφαρμογές. Εάν θέλουμε να υπάρχει διασύνδεση μεταξύ βιομηχανίας και έρευνας, τότε ε, θα μπορέσουμε να επιτύχουμε και απασχόληση και νέα προϊόντα και θα υπάρξουν και περιττέρω προς για να ε, κατασκευάζουμε στην Ευρώπη πράγματα τα οποία τώρα εισάγουμε από εκτός της Ευρώπης και αυτό πρέπει να σταματήσει. Και είναι κάτι που μας ενδιαφέρει και μας συμφέρει όχι μόνο βαρχιπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα σχετικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, ε, βλέπουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν πληρώνονται. Το θέμα αυτό της γραφειοκρατίας πρέπει να αλλάξει διότι για να υπάρξει έρευνα, για να υπάρξει ανάπτυξη και εργασία και απασχόληση θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όσον αφορά τα κράτη-μέλη ε, γενικώ συμφωνώ ότι πρέπει να τα στηρίξουμε αλλά θέλετε ε, την αριστεία χρειάζονται μεν ε, τα κεφάλαια πρέπει να προωθήσουμε τα τελευταία μέλη που εισήλθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μακροπρόθεσμα θα πρέπει να στηριχθούν όλοι για να μπορέσουμε να επιτύχουμε το στόχο μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Προβέρεντε Κάμπος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να επικεντρωθώ στο θέμα των προτεραιοτήτων. Αυτό που κάποιος ονόμασε τις εκλογές μας. Τι εκλογή θα κάνουμε δηλαδή. Είναι πολύ σημαντικό 80 εκατομμύρια δεν μπορεί να μας φτάσουν εφόσον έχουμε τέτοιο πολλαπλασιασμό των στόχων των προγραμμάτων. Αλλά από την άλλη υπάρχουν και περικοπές στα κονδύλια. Πού όμως βρίσκονται αυτά τα προστατευτικά για τις περικοπές μαξιλαράκια που θα μας προστατεύσουν. Ο κύριος Έλερ μίλησε για το κόστος που μπορεί να έχει η ευκαιρία για τα μεγάλα προγράμματα. Νομίζω λοιπόν οι διαπραγματεύσεις για τις περικοπές είναι αυτό που θα καθορίσει το πώς θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα. Δεν μπορεί να σκεφτούμε να μην σκεφτούμε μάλλον τι θα προκύψει από τις χαμένες ευκαιρίες. Αυτό θα πει μείωση του κόστους. Η πιο κοντινή εναλλακτική χρήση βεβαίω είναι μία λύση. Αλλά για τη συζήτηση αυτή, Πρόεδρε, δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Κανένα, καμιά πληροφορία. Δεν ξέρουμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα με τα καταμεονεκτήματα τη κάθε γραμμή του προγράμματο. Προσπαθήσαμε να παρακολουθήσουμε τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσε. Αλλά περιμένουμε και τη μελέτη αντικτύπου το σχετικό έγγραφο για να δούμε τι γίνεται με κάθε γραμμή του όλου προγράμματο. Αυτό θα μα διαφωτίσει πραγματικά και είναι καθοριστική σημασία. Μπορεί το πρόγραμμα να μην είναι βιώσιμο και για το ε, ίδρυμα, το Ινστιτούτο, συγγνώμη, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομία και Τεχνολογία. Επισκέφτηκα την έδρα του Ινστιτούτου. Ε, κονάκον το επισκέφτηκα μαζί με άλλους συναδέλφους και πρέπει να πω ότι στις συζητήσεις που είχαμε το διευθυντή του Ινστιτούτου ήταν πραγματικά εξαιρετική όλη του αντίληψη για το εγχείρημα και ο ενθουσιασμός του. Ήταν ε, πραγματικά κάτι που μας ενέπνευσε. Αλλά όταν επισκέφτηκα την έδρα πρέπει να πω ότι έζησα μια φοβερή απογοήτευση. Όπως ε, λίγο πολύ όταν επισκέφτηκα και ένα κικ. Αυτό το πρόγραμμα τώρα θέλουμε να το δεκαπλασιάσουμε. Είναι πάρα πολύ αυξημένος ο βαθμός κινδύνου. Και εδώ θα συμφωνήσω απολύτως με τον συνάδελφο Λαμπέρ ε, και όλους τους υπόλοιπους που είπαν ότι αυτό το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Ευχαριστούμε κύριο Πρόντι. Ευχαριστώ Πρόεδρε να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Ριέρα Μαντουρέλ για την παρουσίασή της. Είναι ελάχιστος ο χρόνος, οπότε μόνο κάποια προβλήματα μπορούν να τεθούν κάποιοι προβληματισμοί. Ήθελα να σταθώ σε ένα στοιχείο ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, το θέμα της υγείας και για το πώς θα μπορούσε να υπάρξει γονιδιακή θεραπεία μαζί με την εξέταση των δεοντολογικών προβλημάτων, των ηθικών μάλλον προβλημάτων. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει εμβάθυνση και τεχνολογική και επιστημονική για κάτι για ένα τόσο σημαντικό σκέλος του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, το θέμα είναι τι γίνεται με τις μεγάλες ευκαιρίες, αλλά και τη δυνατότητα, λόγου χάρη το γονιδίωμα, να περιγραφεί πλήρως αυτό ενέχει και ένα κίνδυνο. Η γνώση να μην επιτρέψει την πρόοδο. Πώς θέλουμε λοιπόν να προχωρήσουμε στην ε, γονιδιακή αυτή έρευνα. Μπορεί να υπάρχουν εδώ τεράστιες δυνατότητες μείωση κόστους, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Αλλά από την άλλη θα πρέπει να έχουμε βεβαιωθεί ότι αυτού του είδους η έρευνα δεν θα δημιουργήσει προβλήματα, προβλήματα στα επιμέρους άτομα. Διότι το απόρριτο μπορεί να, να είναι ένα θέμα, η εμπιστευτικότητα των στοιχείων. Μπορεί μια γονιδιακή πληροφορία να κατευθύνει λόγου χάρη τις ασφαλίσεις, τις ασφαλίσεις υγείας. Άρα με εδώ πρέπει να γίνει ένας σαφής διαχωρισμός, ορισμός κινδύνου. Μπορεί κάτι να επιβαρύνεται λόγου χάρη από τη συμπεριφορά της τάσης ζωής του ατόμου ή καθορίζεται πλήρως από το ίδιο το γονιδίωμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν εδώ αυτό το δίνω χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ήθελα να σταθώ σε αυτό για να καταλάβουμε και όλα τα υπόλοιπα. Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το δούμε και από τις δύο του όψεις. Από τη μια επιστημονική εξέταση του ζητήματος, επιστημονική εμβάθυνση, αλλά από την άλλη υπάρχει και το θέμα της νοοτροπίας και του πώς ηθικά αντιλαμβανόμαστε το ζήτημα του απορρίπτου και των εμπιστευτικών πληροφοριών. Ευχαριστούμε κύριε Βεβέρ. <clears throat> Ευχαριστώ. Σε δύο λεπτά, όπως και ο κύριος Πρόντι που επικεντρώθηκε σε ένα θέμα, θα επικεντρωθώ και εγώ σε ένα και μοναδικό που με ενδιαφέρει και μας απασχολεί πολύ. Είναι το σκέλος που αφορά το διάστημα. Ένα δις 737 εκατομμύρια ε, προβλέπονται για αυτή την περίοδο με μεγάλα θέματα. Ε, γενικά μας ικανοποιεί καλύπτει την υποστήριξη στην καινοτομία και τις τεχνολογίες που είναι αποφασιστικές για να εξασφαλίσουμε την ευρωπαϊκή ανεξαρτησία και τα συστήματα ε, παρακολούθησης του διαστήματος για να προστατεύουμε τους δορυφόρους μας από τα απόβλητα που περιφέρονται στο διάστημα. Στη σημερινή πρόταση, σε σχέση με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, ε, είναι ο προϋπολογισμός ε, σταθερός, αλλά θα πρέπει να επαγρυπτούμε για να διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα. Και θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας διαβεβαιώσει ότι το πρόγραμμά της θα είναι πλέον πιο φιλόδοξο από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για τις τεχνολογίες διαστημικής μεταφοράς και τη διερεύνηση. Παράδειγμα, λείπει ένα σημείο που θεωρώ θεμελιώδες στους στόχους για το 2020, είναι αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε εντός εισαγωγικών το αηφόρο διάστημα. Δηλαδή πέρα από την παρακολούθηση των αποβλήτων θα πρέπει να προβλέπει και την εξάλληψή του, την πράσινη ανάπτυξη και με ανακύκλωση, βελτιστοποίηση γενικά των ε, διαστημικών αποστολών και παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και μη ρηπογόνου όπως ε, είναι οι ηλιακοί συλλέκτες ε, στο διάστημα σε ό,τι αφορά το GMES για την ε, παρακολούθηση κλιματικής ε, αλλαγής. Υπάρχει αντίστοιχο κεφάλαιο ε, για την προστασία του κλίματος, για τις πρώτες ύλε, αλλά δεν αναφέρεται πουθενά συγκεκριμένο ποσό. Είναι γεγονός ότι επικρατεί εκεί κάποια ανασφάλεια και γενικά για το πρόγραμμα στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές και αυτό παραμένει πρόβλημα. Επίσης, Σημειώνω, όπως και ορισμένοι προλαλήσαντες, ότι το ποσό ε, ε, ειδικά για το Γαλιλαίο επίσης δεν αναφέρεται. Και θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτά τα σημεία. Οι τελευταίες δύο παρεμβάσεις. Κυρία Νίμπλε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη για να μπορέσουμε να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ την κυρία Μαντουρέλ για το εξαιρετικό έγγραφό της που μας έδωσε τη δυνατότητα να δομήσουμε σωστά τη συζήτηση και όλους τους παρεμβαίνοντας μέχρι τώρα. Θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Καταρχήν θεωρώ ότι και η βασική διαμόρφωση του προγράμματος και η δόμησή του ακολουθεί μία γραμμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή ε, ε, Ευρώπη του 2020, ορίζοντας 2020, όπως επίσης και ε, μία διαμόρφωση που προβλέπει πώς θα είναι η καινοτομία και η έρευνα το 2020, ότι προσπαθεί όλα αυτά να τα συγκεράσει σε ένα ενιαίο σύνολο, αυτά θεωρώ ότι είναι πολύ θετικά στοιχεία. Τώρα, σχετικά με την ε, πρόταση του προϋπολογισμού, 80 δισεκατομμύρια δεν είναι το τέλος του κόσμου. Όπως είπε η κυρία Μαντουρέλ πολύ σωστά στο έγγραφό της, ουσιαστικά αν λάβουμε υπόψη όλα τα προγράμματα έχουμε μία αύξηση 6% για τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας και δεν νομίζω ότι είναι το τέλος του κόσμου οπότε δεν ξέρω πόσο ε, σκέφτεται ότι θα μπορέσουμε να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό όταν όλα τα ε, κράτη ε, καλούνται να καλύψουν από το ΑΕΠ τους 3% κάθε χρόνο. Το 2001 είμαστε στο 1,6% και βλέπουμε ότι το 2010 ήμασταν στο 2%. Δηλαδή μία οριακή αύξηση κατά 0,1,4 ίος και αν προχωράμε έτσι δεν ξέρω πότε θα φτάσουμε το 3%. Λοιπόν, δεν ξέρω ε, πώς τα βλέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα τα πετύχει όλα αυτά. Όσον αφορά τους συναδέλφους οι οι οποίοι ε, κατέκριναν την ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία πρέπει να δούμε ε, τι μπορεί να υπάρξει στον προπολογισμό και στο ίτερ για το μέλλον. Είμαι υπέρ ε, της βασικής έρευνας διότι το 2007 ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια και πιστεύω ότι έχει αποτελέσει έναν πυρήνα προωθήσεως στην Ευρώπη και γι' αυτό ε, θα πρέπει στην βασική έρευνα να διπλασιάσουμε τη χρηματοδότηση. Επίσης άλλοι συνάδελφοι ε, ανέφεραν ε, διάφορα θέματα. Πρέπει να δούμε πώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά πιο αποτελεσματικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μας εξηγήσει καλύτερα πώς το σκέφτεται. Επίσης όσον αφορά τα dedicated instrument και τα equity and debt facility και η σχετική πρόταση, τι εννοούν με αυτό. Ε, θα ήθελα να έχω περισσότερες πληροφορίες και γενικώ να δω πώς μπορεί κανείς να εμπλέξει περισσότερο τον ιδιωτικό τομέα πέραν των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διότι αυτά ήταν τα θυμία που είχαμε κατακρίνει στο προηγούμενο πρόγραμμα έρευνας του ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το ζήτημα είναι σημαντικό. Είναι θεμελιώδου σημασία αυτό το ντοσχέ για την ανάπτυξη. Νομίζω λοιπόν ότι αξίζει της προσοχής μας το σύνολο αυτών των προτάσεων, αλλά να επισημάνω το εξής στην εισηγήτρια. Εάν θέλετε να με ακούσετε, ε, είμαι εδώ. Καλό θα ήταν να με ακούσετε. Πολύ θα μου άρεσε. Α, είναι ο Ναι. Εντάξει, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ακούσετε αυτήν την έκκληση, την ισχυρή έκκληση. Μην διστάσετε και μην φοβηθείτε για το για τη χρηματοδότηση του προγράμματος. Ε, η κρίση αυτή έχει γίνει κάτι σαν αλυσίδα που μας έχει, έχει λειτουργήσει ως όριο για να προωθήσουμε νέες πρωτοβουλίες. Όμως, πιστεύω υπάρχει ζήτηση για το πρόγραμμα αυτό και από ιδιώτες. Άρα αυτό θα πει ότι είναι επιτυχημένο το πρόγραμμα και αυτό μπορεί να είναι κάτι που θα κινητοποιήσει και τον κρατικό, τον δημόσιο τομέα. Είναι δηλαδή κάτι που συναρθρώνει τον ιδιωτικό με τον δημόσιο τομέα και τόσα πολλά προβλήματα, όσα πολλά προβλήματα και αν υπάρχουν μπορούμε να τα λύσουμε. Πρέπει λοιπόν να δούμε σε ένα κοινό πλαίσιο τα ιδιωτικά και τα δημόσια κονδύλια. Εκεί θα μπορούσαμε να κάνουμε το λεγόμενο μίξ, ένα μείγμα, ένα συνδυασμό ώστε να υπάρξει ένα σύνολο προτάσεων πιο συγκεκριμένων. Νομίζω λοιπόν ότι καλό είναι να ενδιαφερθούμε για αυτή την σκοπιά γιατί για πολλά ερευνητικά προγράμματα θα υπάρξει περιορισμένη ε, ε, κρατική παρέμβαση και χρηματοδότηση αλλά υπάρχουν και οι εφαρμοσμένες τεχνολογίες και η αγορά και Σίγουρα η βάση όλων αυτών είναι η στηρίξη από τα ερευνητικά ιδρύματα. Αυτό είναι λοιπόν έκκληση που την απευθύνω σε όλους, αλλά σε εσά ιδιαίτερω. Και από την παρουσίασή σας μου φάνηκε ότι έχετε και εσείς ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτό το σημείο. Τελευταία παρατήρηση. Παρατήρηση ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν περιλαμβάνεται πλέον μεταξύ των προτεραιοτήτων. Αυτό οφείλεται στη δική σας παρέμβαση. Είναι μια αμέλεια, περιλαμβάνεται σε κάποιο άλλο πλαίσιο. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριος Σμιτ, Γενικό Διευθυντή για την Έρευνα και την Ανάπτυξη. Well, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πολύ εμ, ζωντανή συζήτηση και εμπλουτιστική. Ευχαριστώ όλους τους παρεμβαίνοντες για τα ενδιαφέροντα σχόλια. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους τέσσερις εισηγητές και τους Σκιώδης και τους ε, υπολείπους βουλευτές που πήραν το λόγο. Ιδιαίτερα επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω την κυρία Μαντουρέλ για το σχέδιο έκθεσης της και τις τεράστιες προσπάθειες που έκανε για να την υποβάλει εγκαίρως. Γιατί πραγματικά ο χρόνος είναι το σημαντικό αυτή τη στιγμή έτσι ώστε να εγκριθεί ταχύτατα η πρόταση. Ε, η έκθεση είναι μια πολύ καλή αφετηρία πιστεύω και χαίρομαι πολύ που ε, είναι θετική ε, απέναντι στον ορίζοντα 2020. Γενικά εγκρίνεται την προσέγγιση, τη δομή, τους στόχους ε, και τη μέθοδό μας και νομίζω ότι είναι ευρία η αντίληψη αυτή στην Επιτροπή σας και φαίνεται και από την έκθεση. Ο κύριος Τσουκαλάς αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο ιστορικό πριν συζητήσουμε τέτοιες προτάσεις, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πού βρίσκεται η Ευρώπη στο παγκόσμιο σκηνικό, σκηνικό συγγνώμη, σε σχέση με τους ανταγωνιστές. Εκπαιδεύουμε σωστούς ερευνητές με αρκετά χρήματα, είμαστε ισχυροί στην έρευνα, στην καινοτομία. Τι μας λείπει. Πριν καταθέσουμε την πρότασή μας, κάναμε εκ των προτέρων βαθύτατη συζήτηση με ε, φορείς καινοτομίας. Ε, με χαρά να σας δώσουμε τα στοιχεία γραπτός ή προφορικός, γιατί πριν καταθέσουμε αυτή την πρόταση, ορίζον 2020, κάναμε μια βαθύτατη ανάλυση για το πού βρίσκεται η Ευρώπη στο παγκόσμιο σκηνικό. Η κυρία Νίμπλερ το ανέφερε ότι ακόμα δεν είμαστε εκεί που θα έπρεπε. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων είπαν ότι το 2010 θα έπρεπε το 3% να πηγαίνει στην έρευνα. Έχουμε κολλήσει στο 2%. Δεν έχουμε αρκετούς ερευνητές ε, στους χίλιους εργαζομένους, ούτε εξάγουμε πολλά προϊόντα υψηλής ε, τεχνολογίας, ούτε διπλώματα ευρυσιτεχνίας έχουμε που θα οφείλαμε. Υπάρχει πρόβλημα συνεργασίας ε, της βιομηχανίας με τα πανεπιστήμια. Ακριβώς εντοπίζοντας τις δυσκολίες, εκεί εστιάσαμε και την πρότασή μας. Σε ό,τι αφορά τώρα ορισμένα στοιχεία που αναφέρθηκαν ε, κατά τη διάρκεια της συζήτησης και τα λέει και η έκθεση κυρίας Μαντουρέλ. Πρώτα απ' όλα, ο προπολογισμό. Ο κύριος Λαμπέρτς αλλά και άλλοι αναλύσατε τη σημασία των μέτρων αύξηση τη οικονομία. Δεν μπορεί η Ευρώπη να οικοδομηθεί στο μέλλον βασιζόμενη στη δημοσιονομική πειθαρχία και στη λιτότητα. Θα πρέπει να ενταθεί η ανάπτυξη με συγκεκριμένες δραστηριότητες και αμέσως πάει το μυαλό μα εκεί στην καινοτομία και στην έρευνα. Εξού και η έκθεση ΟΝΤΗ, τα 100 δισεκατομμύρια που ζητήσατε και θεωρήσατε ότι πρέπει να είναι ο μελλοντικό προπολογισμό του ορίζοντα 2020 είναι ένα ισχυρό μήνυμα και προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προ το Συμβούλιο. Γιατί σε τελική ανάλυση ο προπολογισμό είναι το στοιχείο που ακριβώ θα κάνει τη διαφορά. Σε ό,τι αφορά ακριβώ λοιπόν τον προπολογισμό και την κατανομή του, Είδα ότι πολλοί από εσά υποστηρίζετε πολύ το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Συμβούλιο και κυρία Νίπλερ, ευχαριστούμε έχετε προηγούμενη εμπειρία από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, αλλά και άλλοι, όχι μόνο η κυρία Η κυρία Μαντουρέλ εντόπισε το πρόγραμμα Marie Curie ότι υποχρηματοδοτείται. Αυτό είναι ένα θέμα που αναφέρεται ρητά στην έκθεσή σας, όπως και άλλοι τομείς ε, που χρειάζονται ε, περισσότερη πρικοδότηση από πλευράς προϋπολογισμού. Η μόχλευση είναι ένα σημαντικό στοιχείο και πολλοί από εσά υπογραμμίσατε τη σημασία να χρησιμοποιείτε ο προπολογισμό του προγράμματος αυτού ακριβώς προς το συγκεκριμένο σκοπό. Τα χρηματοδοτικά μέσα που προτείνουμε, ε, equity και debt, εξορισμού ε, είναι ε, πρόσφορα. Ο κύριος Έλερ γνωρίζει καλά το μηχανισμό και σύμφωνα με ε, ανεξάρτητες ε, πηγές έχει 15πλάσια ε, απόδοση. Αυτό το λένε ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες. Το έκανε μια πρώην συνάδελφό σας, η Έρικα Μαν. Πριν από λίγους μήνες ήρθε και κατέθεσε την έκθεσή της Οπότε τα χρηματοοικονομικά μέσα που είναι μέσα δανειοδότησης, εξορισμού, είναι πρώτη τάξεως μέσα και προσφέρονται για μόχλευση. Υπάρχουν όμως και άλλα, όπως είναι η ΣΔΙΤ, οι κοινέ τεχνολογικέ προσπάθειες. επίση εξορισμού είναι καλά μέσα για να δοθεί μια όθηση και στη βιομηχανία. Το κάναμε, νομίζω, με τρόπο αρκετά επιτυχή. Θυμάμαι πρόσφατα, ε, η κυρία Καρβάλιο είχε διοργανώσει ε, μια ε, ακρόαση για τα τζέτης και πόσο σημαντικά είναι. Πραγματικά αυτό το έχουμε υπόψη μας και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα Horizon 2020. Τώρα, ακούστηκαν οι κοινωνικές επιστήμες και στην έκθεση Ματουρέλ τίθεται το ερώτημα γιατί συνδέονται με την ασφάλεια αυτές. Δεν θα πρέπει να είναι χωριστή προτεραιότητα. Η δική μας προσέγγιση σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές επιστήμες ήταν η εξής. καταρχάν θέλουμε να ε, μπουν ε, στη βασική προσπάθεια ε, στο mainstream, δηλαδή ο, ο πληθυσμός γυράσκει, έχουμε θέματα ενεργειακής ασφάλειας, επιστημιστικής ασφάλειας, οι κοινωνικές επιστήμες μπορούν να συνεισφέρουν. Και πραγματικά θα πρέπει να έχουμε πολλά χρήματα και για τις επιστήμες αυτές, τις θεωρητικές και κοινωνικές. Αλλά ε, είναι στην ίδια επικεφαλίδα και στον ίδιο τίτλο με την ασφάλεια. Όταν μιλούμε για τρομοκρατία, για ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, για την ανασφάλεια που ζουν οι πολίτες, ε, εδώ έχει να κάνει με τις κοινωνικές επιστήμες που αν δεν παρέχουν τη λύση, παρέχουν τουλάχιστον την εξήγηση. Τα αίτια της τρομοκρατίας θα πρέπει να τα κοιτάξουμε και από πλευράς κοινωνικής και από πλευράς ε, ανθρωπιστικής. Εδώ λοιπόν έρχονται να ενταχθούν οι κοινωνικές και θεωρητικές επιστήμες. Άρα έχει νόημα αυτή η διάρθρωση που βάλαμε στο ίδιο κεφάλαιο τα θέματα αυτά των κοινωνικών επιστημών σε στενή διασύνδεση με τις διάφορες ε, ενότητες. Ε, τώρα, έρχομαι στο τίτλο των στόχων. Υπάρχει μια καινοτομία εδώ. Οι δείκτες, οι δείκτες τους έχουμε εντοπίσει και μετά θα μας βοηθήσουν εκ των υστέρων να εκτιμήσουμε τον αντίκτυπο του Horizon 2020. Αυτό είναι καινούριο. Δεν το είχαμε σε προηγούμενα προγράμματα και βλέπετε για πρώτη φορά το Κοινοβούλιο, και το αναφέρει πανελιμένα ε, ε, έχουμε ένα κατάλογο πλέον δικτών για να μας βοηθήσουν μετά να κάνουμε τη μελέτη αντικτύπου. Βεβαίω ήδη έχουμε κάνει εκ των προτέρων κάποια εκτίμηση για τον αντίκτυπο του ορίζον 2020, ποιε και πόσε θέσει απασχόλησης θα δημιουργηθούν, ε, ακόμα και αύξηση του ΑΕΠ. Έχουμε κάνει αυτές τις προβολέ, υπάρχουν τα στοιχεία στη διάθεσή σα. Είναι σημαντικό να δείξουμε την προστιθέμενη αξία ακριβώ να πιάνει τόπο το κάθε ευρώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο που δαπανάτε. Η κυρία Τζόρνταν, ο κύριος Έλερ και πολλοί άλλοι μίλησαν για την αριστεία και ε, την πορεία και μια κλίμακα προς την αριστεία. Ο ορίζον 2020 δεν απευθύνεται σε ένα περιορισμένο αριθμό κρατών αλλά και στα 27 κράτη μπορούν να συμμετέχουν και να επωφεληθούν από αυτό. Αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ κρίσιμο, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και κάναμε και προτάσεις. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε αφενός ότι εντός των διαρθρωτικών ταμείων υπάρχουν αρκετοί πόροι οικονομικοί διαθέσιμοι έτσι ώστε οι λιγότερο επιτυγμένες περιφέρειες της Ευρώπης να αναπτύσσουν δυνατότητες έρευνας και καινοτομίας. Τα ποσά είναι 60 με 80 δις εκατομμύρια ευρώ την επόμενη επταετία ας πούμε για εξυγχρονισμό πανεπιστημίων, για υλικοτεχνικό εξοπλισμό, υποδομές, ε, συστήματα κλιβάνων ας πούμε, τεχνολογίας, ε, μεταφοράς τεχνολογίας για να μπορέσουν οι περιφέρειες αυτές να εξυγχρονίσουν τις υποδομές του και να ξαναχτίσουν τη δυνατότητα για καινοτομίες. Ας πούμε, Ιρλανδία, Ισπανία, στο παρελθόν και η Ελλάδα ε, το συζητήσαμε την περασμένη φορά για την Κρήτη. Ε, χρησιμοποιούν τα χρήματα αυτά με τρόπο ευφυή και πραγματικά δημιούργησαν έτσι μια κλίμακα προς την αριστεία. Αυτό όμως δεν αφορά μόνο τα διαρθρωτικά ταμεία. Για να διευρυνθεί η συμμετοχή προβλέπουμε πάντα στο ορίζον 2020 ε, διασύνδεση, αδελφοποίηση, έδρες συγκεκριμένε έρα, έτσι ώστε έχουμε προβλέψει πολλά για να εποφελείται το σύνολο της Ευρώπης και όχι ένα μικρό τμήμα. Επιευκαιρία να σας πω ότι επειδή συνδέεται με τα διαρθρωτικά ταμεία ε, ορίζον 2020 και αυτό σας ενδιαφέρει πολύ, συνεννοηθήκαμε με τους συναδέλφους της ε, Γενικής Διεύθυνσης για τα περιφερειακά ζητήματα να κάνουμε ένα κοινό έγγραφο και να το υποβάλουμε σε εσά για να δείτε πόσο στενή είναι η συνεργασία μας για να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν πραγματικά αυτές οι συνέργειες και μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτή την κλίμακα προς την αριστεία. Ένα πολύ θετικό στοιχείο εδώ είναι ότι οι συνάδελφοι της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακών ε, Θεμάτων μας ζήτησαν να συμμετέχουμε και στη διαπραγμάτευση, στις ομάδες που θα διαπραγματευτούν ε, τι συμβάσεις εταιρικές που αναφέρθηκε ο κύριος ε, Φανίστερόι για να υπάρξει η ευφυής εξειδίκευση. Συνεργάζονται λοιπόν ε, με τρόπο υπαδειγματικό οι δύο γενικές διευθύνσεις και το έγγραφο που εκπονούμε από κοινού πολύ σύντομα θα σας υποβληθεί. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε μερικά ζητήματα ακόμα. Απλούστευση. Όπως γνωρίζει η κυρία Καρβάλιο, τα περίφημα 67 μέτρα της απλούστευσης δεν είναι ακριβώς στο προσκεφάλι μου, ε, αλλά είναι πολύ κοντά ε, και ε, με απασχολούν. Είναι τρία τα βασικά μέτρα που πρέπει να συζητήσουμε, τα χρονοδιαγράμματα, το πλήρες οικονομικό κόστος και ένα ακόμα, όχι βέβαια το λιγότερο σημαντικό είναι ε, πότε ε, θα γίνονται οι συμβάσεις. Δηλαδή θα πρέπει άπαξ και διαπαντός να πατάξουμε αυτό το τέρας της γραφειοκρατίας. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας και αυτά τα 67 μέτρα που προτείνετε είναι πραγματικά τα σωστά βήματα για την απλούστευση. Επίσης ελπίζουμε να έχει αντίστοιχη προσέγγιση και το Συμβούλιο Πάντως αισιοδοξώ ότι και τα κράτη-μέλη θέλουν να πατάξουν αυτό το τέρας γραφειοκρατίας και να το ε, δαμάσουν και να το βάλουν ξανά στο κλουβί του. Ε, άλλα θέματα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στον ορίζοντα 2020 δίνουμε πολλά χρήματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κοιτάξτε, εάν υπολογίσετε τα χρήματα που καταρχήν διατίθενται ε, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι 8,6 δισεκατομμύρια. Είναι πολλά τα λεφτά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. SPIR είναι το νέο σύστημα που έχουμε αντιγράψει από τις Ηνωμένε Πολιτείε για την ενίσχυση των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα βεβαιωθούμε ότι θα είναι κομμένο και ραμμένο στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Να είστε βέβαιοι λοιπόν ότι θα είναι οι κύριοι δικαιούχοι του προγράμματος Horizon 2020. Στη συνέχεια να πω και δύο λόγια για το EIT, το Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο. Κάτι ρωτάει ο κύριος Σέλερ εκτός μικροφών. Α, πώς ορίζεται η μικρομεσαία επιχείρηση. Μα υπάρχει επίσημος ορισμός στα ευρωπαϊκά προγράμματα των μικρομεσαίων. Υπάρχει ένας ορισμός τον οποίο τηρούμε. Ε, για να έχουν πρόσβαση ε, στο νέο σύστημα, το ζήτησε η κυρία Νίμπλερ, οι οροφές να είναι πολύ χαμηλότερες. Δηλαδή τα δάνεια ανά έργα μπορεί να είναι πολύ χαμηλότερα και αυτό είναι μια προσέγγιση νομίζω φιλική προς τις μικρομεσαίες. Για το Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο που σας έλεγα είναι μια έννοια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διότι ε, ενώνει αυτό το περίφημο τρίγωνο. Είναι τεράστιο το δυναμικό, η δυνατότητα και η κίξη οι κοινότητες ε, γνώσης και καινοτομίας ζητούμε αύξηση του προπολογισμού γιατί πραγματικά θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Υπάρχουν και συνάδελφοι από άλλη γενική διεύθυνση που αν θέλετε μπορούν να σας ενημερώσουν. Ε, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και πολιτιστική κληρονομιά, όχι. Καλύπτεται θα στείλω στον συνάδελφό σας που αποχώρησε ε, τις αντίστοιχες προτάσεις. Βεβαίως είναι σημαντική πολιτιστική κληρονομιά και σε καμία περίπτωση δεν θα την ξεχνούσαμε. Ένα τελευταίο, χωρί δεν είναι το λιγότερο σημαντικό, μερικά λόγια για την καινοτομία. Ο Δόκτωρ Έλερ και κάποιοι άλλοι τα ανέφεραν και η κυρία Μαντουρέλ το λέει στην έκθεσή τη. Η καινοτομία βεβαίω δεν περιορίζεται αυστηρά στον πυλώνα τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα. Διαπερνά το σύνολο. Αν δείτε τη θεμελιώδη έρευνα, τον πυλώνα της αριστείας, υπάρχει και εκεί ακόμα καινοτομία. Συγκεκριμένα μέτρα για να περάσουν τα αποτελέσματα της θεμελιώδους έρευνας στην αγορά. Επίση και προκλήσεις για την κοινωνία. Δεν θέλουμε μόνο να αναπτύξουμε την έρευνα, αλλά και την καινοτομία και τα αποτελέσματα της έρευνας να βγουν στην αγορά για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Η καινοτομία είναι πραγματικά ε, εκ των ονουκάνευ. Προτείνουμε στην υγεία, στην ενέργεια, ε, σε θέματα τροφίμων, μεταφορών, επιδείξεις, έτσι ώστε να υπάρχουν ε, ευρύτατες προσπάθειες η απόδειξη των ενιών proof of concepts και τα λοιπά να φτάνουν και στην αγορά. Και βεβαίως η καινοτομία στον τελευταίο πυλώνα που είναι η βιομηχανική ηγεσία. Η καινοτομία δεν είναι κάτι το οποίο αφορά ένα και μόνο πυλώνα, αφορά το σύνολο γιατί περί αυτής πρόκειται. Ορίζον 2020 ε, αφορά την υλοποίηση, αφορά τα αποτελέσματα της έρευνας να φτάνουν στην αγορά, να είναι ολοκληρωμένη προσπάθεια έρευνας και καινοτομίας, να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα τη βιομηχανία μα και να βεβαιωθούμε ότι για τους πολίτες αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις κοινωνίας. Συγγνώμη που μακρηγόρησα τόσο πολύ και σας ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστούμε τον Γενικό Διευθυντή για τις αποκρίσεις του. Έχουμε ξεφύγει λίγο από το χρόνο που προβληπόταν. Όμως να θυμίσω στους συναδέλφους ότι στις 20 Μαρτίου 2012 έχουμε μια ακρόαση. Εάν κάποιος συνάδελφος θέλει κάτι να προσθέσει, συντομότατα για λίγα λεπτά. Κύριο Σέλερ. Δεν θέλω να σχολιάσω, αλλά ευχαρίστως θα ήθελα να αναφερθώ στο χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή υπήρξε μία πρόταση να, η προθεσμία για τις τροπολογίες να είναι για τις 7 Ιουνίου και η συζήτηση του σχεδίου της εκθέσεως τέλος Μαΐου. Αλλά αν δούμε ρεαλιστικά πόσος φόρτος εργασίας μας περιμένει, νομίζω ότι δεν συνάδει με τον χρόνο ο οποίος θα διατεθεί από την κατάθεση του σχεδίου ο εκθέσεως μέχρι την υποβολή των τροπολογιών και πιστεύω ότι οι τροπολογίες θα έπρεπε να έχουν προθεσμία μέχρι τον Ιούλιο και να ξανασυζητηθεί μετά το καλοκαίρι καλοκαίρι διότι αν έχουμε 700 ή 800 ή 1000 τροπολογίες χρειάζεται κανείς χρόνο να τις διαβάσει όλες και θα ήθελα να υπάρξει συμφωνία μεταξύ μας διότι διαφορετικά από την πείρα μας δεν είναι δυνατόν έχοντας, ανατρέχοντας στο σχέδιο πλαίσιο 7 να προχωρήσουμε με τέτοιους ρυθμούς. Κυρία Μαντουρέλ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Το θέμα του χρονοδιαγράμματος που μας προτείνει ο κύριος Σέλερ μπορούμε να το συζητήσουμε την επόμενη φορά που θα είναι παρόντες όλοι οι ηγητές και οι σκιώδεις. Καταρχήν είναι προσανατολιστικό αυτό, δεν έχω κανένα πρόβλημα ε, δεκτικό το χρονοδιάγραμμα. Δεν μπορώ να σχολιάσω όσα υπόθηκαν, απλώ να ευχαριστήσω στο ένα λεπτό που έχω του συναδέλφου για τα σχόλιά του, όλου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενημέρωση και για την απάντηση στις ερωτήσεις που κάναμε. Όλα ήταν πολύ ενδιαφέροντα και πάρα πολύ εύστοχα. Εγώ πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχω περισσότερες ερωτήσεις ακόμα από απαντήσεις. Οπότε θεωρώ πολύ χρήσιμα τα όσα άκουσα. Θα συνεργαστώ με όλους τους συναδέλφους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να φτάσουμε σε συμφωνίες. μόνο πώς αλλιώς θα μπορούσαμε άλλωστε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε συνάδελφος Καρβάλιου. Κανείς άλλος. Ωραία. Ολοκληρώσαμε τις εργασίες μας που για το Προεδρείο βέβαια και κάποιους συναδέλφους θα συνεχιστούν με τις συνεδρίες των συντονιστών. Σας ευχαριστούμε. Θα τα πούμε αύριο το πρωί.